ανακοίνωσε την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του κυρίου Πάλμερ από τις 3 Οκτωβρίου του 2017 και αντικαθιστά την κυρία Βίλμοτ. Το Κοινοβούλιο σημειώνει την εκλογή του. Καλώς ήλθατε συνάδελφε και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να σεβαστείτε όλες τις προϋποθέσεις του κανονισμού. Μετά από